αναπτυσσόμενες χώρες. Το λόγο έχει η κυρία Λίντα Μακάβαν, συντάκτης της ερώτησης. Thank you, Mr. President. And, um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας είχαν σαφείς στόχους μεταξύ των οποίων την εξάλληψη της ε, ακραίας ένδυας και τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά παρόλα αυτά ο αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν και υποστήριζονται είναι απαράδεκτα υψηλός. Το ψήφισμα αυτό έχει στόχο να καταστήσει αυτό το ζήτημα πρώτης προτεραιότητας στην συλλογική μας δράση στο πλαίσιο μετά το 2015. Ο υποστηρισμός είναι τεράστια πρόκληση, αναπτυξιακή. Ο ΠΟΗ λέει πως ε, ο υποσυτισμός ε, προφανώς ε, συνεισφέρει κατά πολύ στην παιδική θνησιμότητα και είναι η αιτία του 35% των παιδικών ασθενειών κάτω των 5 ετών. Και βεβαίως είναι η αρχή ενός φαύλου κύκλου που έχει μετά επιπτώσεις και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Γι' αυτό η καταπολέμηση του υποσυτισμού πρέπει να παραμείνει κύριος στόχος στην ατζέντα μετά το 2015. Το ψηφίσαμε αυτό την Τρίτη και είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο σχέδιο εγγράφου της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ, ο στόχος 2 περιέχει έναν στόχο να τελειώσει ο υποστησμός μέχρι το 2035 και μέχρι το 2020 να ε, επιτευχθεί ένας στόχος για την ελληπή σωματική ανάπτυξη των ε, παιδιών. Μέχρι το 2025 αυτό. Αυτό σημαίνει να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που δεν αναπτύσσονται σωστά κατά 70 εκατομμύρια μέχρι το 2025 συνάδελφοι. Στην έκθεση ΣΤΙΕΡ, την Τρίτη το Κοινοβούλιο υπερψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία να στηρίξει αυτόν τον στόχο και πάει παραπέρα και ζητάει την πλήρη εξάλληψη της πείνας μέχρι το 2025. Ζητάει αηφόρο γεωργία και να αναγνωριστούν ειδικά οι ανάγκες των γυναικών γεωργών. Τι ζητάμε λοιπόν από την Κομισιόν και γιατί ζητήσαμε αυτή τη συζήτηση. Χρειάζεται τώρα ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το πώς εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου και πώς θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς μας εταίρους. Οι υπηρεσίες της ε, Κομισιόν ε, επεξεργάζονται ένα σχετικό σχέδιο. Θέλω να μας ενημερώσουν λοιπόν και να μας πούν πότε θα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα και πώς θα έχουμε συντονισμό και εντός της Κομισιόν και με τους διεθνείς εταίρους. Η μείωση της παιδικής, του παιδικού υποστηρισμού είναι δυνατή, αλλά απαιτούνται πόροι, συντονισμός και πολιτική βούληση. Αυτή την εβδομάδα είχαμε την 25η επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού η αντιμετώπιση του υποσυτισμού τα επόμενα 15-20 χρόνια θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά έτσι ώστε το κάθε παιδί να έχει το βασικό δικαίωμα που θα του δώσει την ευκαιρία για μια αξιοπρεπή ζωή. Σας ευχαριστώ. Το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής έχει ο Επίτροπος κ. Χρήστος Τηλιανίδης. Chair, honorable member. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, από πλευράς του Επιτρόπου του κ. Νίμιτσα θα εδώ και να ευχαριστήσω την κυρία Μακαβάνη για το, την προφορική αυτή που είναι τόσο εύστοχη και μας υπενθυμίζει το ότι ο υποσυντισμός δεν είναι μόνο μια υπαρκτή ανθρώπινη τραγωδία αλλά είναι και οικονομικό ζήτημα το οποίο αποτελεί φραγμό στον δρόμο προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να σας τονίσω το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρως δεσμευτεί ούτως ώστε να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση και τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναδειχθεί ως βασικός ε, παράγον για την καταπολέμηση της ε, του υποσυντισμού και γιατί πρόκειται για σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας για την ανάπτυξη. Το 2013 είχαμε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την βοήθεια ε, για την διατροφή και είπαμε ότι έχει δημιουργηθεί μια στρατηγική με στοχος πρωτα πρώτα-πρώτα να μην έχουμε διασπάθηση των ε, τροφίμων και να βοηθούν τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 5. Επίσης, έχει επεξεργαστεί δύο προγράμματα δράσης η Επιτροπή. Το ένα αφορά τον ε, υποσυδισμό και επίσης το να μην ε, γίνεται σπατάλη των τροφίμων και επίση ο άλλο άξονα είναι το να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα για τα 3,5 δις τα οποία έχουν δεσμευθεί ούτω ώστε να βοηθούν τα παιδιά κάτω από τα 5. Και αυτό το πρόγραμμα δράσης δεν προβλέπει μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Επίσης υπάρχει λογοδοσία και θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για την, ε, ε, για την υπόθεση του υποσυτισμού και αυτά είναι οι πυλώνες του προγράμματος δράσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τέτοια παρέμβαση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, άμεσες αιτίες του υποσυτισμού, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται επίσης να αντιμετωπίσουμε τις πιο άμεσες αιτήσεις που πιέζουν, οπότε και θα πρέπει η σωστή διατροφή να ενταχθεί και σε άλλες πολιτικές μας όπως η γεωργία, η παιδεία, η πολιτική για το νερό και γι' αυτό και προχωρούμε όσον αφορά το πρόγραμμα και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε δεσμεύσει 3,1 δις ευρώ για αυτήν την ε, παρέμβαση που θα αφορά τη διατροφή. Αυτό θα γίνει βασικά μέσω της ε, γεωργίας. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης για τη διατροφή. Πάντως για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση πρόκειται να δούμε και να αξιολογήσουμε τι επιπτώσεις και αποτελεσματικό θα έχει το πρόγραμμα και επί τη βάση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών μας θα αποφασίσουμε κατά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το 2017. Να δούμε πώς θα επανακατευθύνουμε κάποιους πόρους, ούτως ώστε ενδεχομένως να βελτιώσουμε τις επιδόσεις κάποιων ε, δράσεων και να μπορέσουμε να πετύχουμε μέχρι το 2025 τους στόχους μας. Οπότε, εν ώψη αυτών των προκλήσεων δεν είναι δυνατόν να δουλέψουμε μόνοι. Προτιθέμεθα στο να επισημαίνουμε σε όλα τα διεθνή φόρα τους κινδύνους από τον υποσυντισμό. Και... Έχουμε 54 χώρες οι οποίες έχουν ασχοληθεί με αυτό το όραμα, αυτό το πρόγραμμα που λέγεται ΣΑΝ και εκτός από τη διεθνή κοινότητα θα συνεχίσουμε και με τον ε, ΦΑΟ και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγεία τη συνεργασία μας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και σε μια διεθνή διάσκεψη για να μπορέσουμε αυτή η πολιτική όθηση για την υπόθεση διατροφή να συνεχιστεί. Αλλά και σε επίπεδο χωρών έχουμε εφαρμόσει την αρχή του να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με το πρόγραμμα μας για την περίοδο 2014-2020. Αυτή την περίοδο προγραμματισμού. Και, τελευταίο αλλά σημαντικό, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και ανταλλαγή εμπειριών. Εν κατακλείδη. Γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του υποσυντισμού απαιτεί συνδυασμένε προσπάθειε σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίω και χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για την υπόθεση αυτή. Σα ευχαριστώ για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα περνούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Ζάμπορσκα, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους, ε, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την πρόεδρο, τη Λίντα Μακέβαν, που ανέλαβε την ε, εισήγηση για το έγγραφο το οποίο εγκρίθηκε στην περασμένη θητεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για την συνεργασία διότι ε, μέσω των ε, τροπολογιών βελτιώθηκε το κείμενο και ευχαριστώ και όλους τους συνάδελφους που ε, βοήθησαν από όλες τις πολιτικές ομάδες. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ψηφίσαμε για το έγγραφο το οποίο θα μας λέει τι θα γίνει μετά από το 2015 με τους στόχους της χιλιετίας. Ο υποσυτισμός είναι περίπλοκο πρόβλημα και αποτελεί βάρος για ολόκληρη την κοινωνία. Πρόκειται για βάρος, διότι με τον υποσυτισμό παραβιάζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή για τα παιδιά που ζουν πεινασμένα. Κάθε λεπτό αρκετά παιδιά πεθαίνουν και αυτό όχι μόνο ε, επειδή ε, είναι άρρωστα ή επειδή έχει πόλεμο στις χώρες τους, αλλά επειδή πεινάνε και... Μπορεί επίσης να αναπτύξουν άλλες ασθένειες ακριβώς επειδή ε, αν επιβιώσουν, επειδή ε, πέρασαν ε, πείνα σε νεαρή ηλικία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε με άλλους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργασία με άλλους οργανισμούς που ε, ασχολούνται με, τις, ε, με τα τρόφιμα όπως η ΦΑΟ. Θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η συνεργασία. Γνωρίζω ότι είπε ο ε, Επίτροπο στη διάρκεια της ακρόσης ότι θα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο τη φτώχεια και την πείνα παρά τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Πάντα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τέσσερα λεπτά η κυρία Πατρίτσια Τόια. Σα ευχαριστώ. Αγαπητέ Επίτροπε, καλωσορίσατε. Θα ήθελα να σα πω ότι αυτή η επαφή στην, σήμερα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πρόκειται για δραματική πραγματικότητα την οποία ε, ε στην ουσία τη δεχόμαστε λες και, ήταν αναπόφευκτη, ε, λες και δεν μπορούσε να αποφευτεί. Ε, είναι πραγματικότητες όμως τραγικές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε ποια είναι τα μέσα που θα έπρεπε να

Ε, χρησιμοποιήσουμε και να το βάλουμε σε εφαρμογή. Γνωρίζουμε τα αίτια αυτών των φαινομένων και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε επίσης. Δεν είναι αναπόφευκτες αυτές οι καταστροφές ε, και πρέπει να αναλάβουμε αυτές τις τεράστιες ευθύνες. Να καταλάβουμε ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί είναι δυνατόν να γίνει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να βάλουμε σε ε, εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα και στο κατάλληλο βαθμό. Ο υποσυτισμός των παιδιών παίρνει μορφές πιο κρυφές, η κρυφή πείνα που είναι λιγότερο προφανής και λιγότερο συνταρακτικές εικόνα που φτάνει στα μάτια μας μέσω των ε, ΜΚΟ, των φορέων ε, διεθνούς συνεργασίας, που είναι όμως επίσης αρνητικές και επιβλαβείς για την ανάπτυξη των παιδιών. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο της κρυφής πείνας, εντάσσεται σε αυτά που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς κινητοποιούμε θα πολύ αυτές τις μέρες με ανανεωμένη δύναμη, ε, ακριβώς επειδή ε, έχουν περάσει και 25 χρόνια από τη δήλωση για τα δικαιώματα του παιδιού και θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής Λίντα Μακέβεν και τους συναδέλφους ε, Σκιώδης ε, ε, γιατί θέλουμε με αυτήν την πρόταση να πούμε ότι η δική μας δέσμευση υπάρχει όχι μόνο της Επιτροπής ΕΝΤΕΒΕ αλλά ολόκληρου του Κοινοβουλίου και ζητάμε από τον Επίτροπο να κάνει αυτό το βήμα μπροστά. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν θα πρέπει και το λέω και εγώ ίδια δεν θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να εορτάσουμε εάν δεν ε, συνοδεύσουμε από συγκεκριμένο δέσμευση. Εσείς μιλήσατε για στοιχεία και για συγκεκριμένα νούμερα, αλλά και συγκεκριμένη δέσμευση που αφορά την αποτελεσματικότητα. Οι πόροι που απευθύνονται στην ε, διεθνή ανάπτυξη δεν χρησιμοποιούνται πάντα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εδώ όμως δεν μπορούμε να χάσουμε πια τίποτα. Ε, πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητά μας, να δούμε τι συμβαίνει με τα προγράμματά μας. Αυτές τις δημεύσεις νομίζω θα πρέπει να τις αναλάβουμε εκ νέου. Με, με, με ανανεωμένο στένος μιλήσατε για την ανάγκη μιας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας για να δούμε πώς θα προγραμματιστούν εκ νέου οι παρεμβάσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να έχετε σε αυτή τη διαδικασία μια πολύ στενή επαφή με το Κοινοβούλιο γιατί θα δείτε ότι έχουμε μεγάλες, ε, πολλά προσόντα, πολύ πάθος και μεγάλο η βούληση για συνεργασία ώστε να ε, γίνουν πιο αποτελεσματικά τα πράγματα. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, πολλά πράγματα. Τα ανάφερε η Λίντα Μακάβαν και εσείς και η Κομισιόν θα πρέπει να είναι περήφανη που συνέβαλε. Όμως επανέρχεται αυτό το φαινόμενο σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές και σε μέρη που δεν υπήρχε λόγω της κρίσης της οικονομικής, λόγω της κερδοσκοπίας, ε, στις τιμές των τροφίμων των βασικών τροφίμων. Ε, οπότε σας ζητάμε να ε, μπορέσετε να, μαζί με τους συνεργάτες να βρείτε μια πολιτική πιο οριζόντια για κάθε πεδίο ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τα αίτια κάποιων από αυτά τα φαινόμενα τα οποία ίσως να βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς ας πούμε με διαφορετική γεωργική πολιτική, διαφορετική εμπορική πολιτική, διαφορετική οικονομική πολιτική. Αυτό το φαινόμενο της κερδοσκοπίας για τα τρόφιμα είναι κάτι το αβάσταχτο για την κοινή γνώμη αυτού του Κοινοβουλίου. Ε, Τέλος, είδαμε όλοι διαβάζοντας και ενημερωνόμενοι, όχι μόνο με αυτή την ευκαιρία, αλλά γενικά για τη δουλειά μας, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας κάνουν πραγματικά να τρέμω. Οι γυναίκες ε, το 80% των τροφών ε, παράγουν στι αναπτυσσόμενες χώρε, και είναι το 60% αυτών που, είναι, ε, που υποφέρουν από υποσυτισμό. Α κάνουμε πολιτική και για τι γυναίκε που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ανάπτυξη σε πολλέ χώρε, όχι μόνο στη Δύση την οποία γνωρίζουμε. Εκ μέρου τη ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Γιάκεβιτς για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, προχτές ο Πάπας είπε πως δεν μπορούμε να δεχόμαστε εκατομμύρια άνθρωποι να πεθαίνουν από την πείνα και να πετάμε τόνους φαγητά από το τραπέζι μας. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ, 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τρόφιμα καταστρέφονται κάθε χρόνο καμία δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καμία χρηματοδότηση για τον υποσυτισμό δεν θα είναι επιτυχής εάν δεν αλλάξουμε τις πρακτικές των ε, κατασκευαστών ε, τροφίμων. Γιατί συζητάμε αυτό όταν μπορεί ακόμα ο κόσμος, ε, κάποιοι δηλαδή, να κερδοσκοπούν με τα τρόφιμα πετώντας τόνους φαγητά για να μην πέσουν οι τιμές. Και μετά τιμωρούνται οι καταναλωτές με επιπλέον φόρους. Πρέπει λοιπόν να... Και μετά μας λέτε εδώ πέρα πως πρέπει να προωθήσουμε τον ρόλο των γυναικών και την ισότητα. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε την αλήθεια. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν σε αυτά τα οποία κάνουν οι βιομηχανίες τροφίμων. Πρέπει να αναλάβουμε σοβαρή δράση ξεκινώντας με την αλλαγή των κανονισμών μας που βλάπτουν τις προσπάθειες που ε, κάνουν οι πιο αδύναμοι. Κύριε Επίτροπε, πείτε μας συγκεκριμένα τι θα κάνετε για να αλλάξουν οι σχετικοί κανονισμοί. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, ο κύριος Λουί Μισελ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο κόσμος βρίσκεται ενώπιν μιας σιωπηρής κρίσης που σαρώνει παντού και προς αυτό το πρόβλημα θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δει τι θα γίνει με αυτή την μάστιγα, την πολιτική, την οικονομική και που αφορά και την ανάπτυξη και που απαιτεί συντονισμό και λογική προσέγγιση. Οπότε είναι και θέμα ηθικό το οποίο δημιουργεί επίσης ε, παραπλευρές οικονομικές συνέπειες. Είπαμε ότι έχουμε ότι έχουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία υποσυτίζονται και ότι έχουμε τη, δεδομένα το ότι ο πρώτος καιρός της ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικός για τα παιδιά και έχουμε αυτή την διατροφική κρίση στο Σαχέλ και στην υποσεχάρια Αφρική. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του κακού. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε αυτό το θέμα από το θέμα της διατροφικής αυτάργειας και θα ήθελα να σας πω μια που έχω εμπιστοσύνη σε εσά στο ότι θα πρέπει όπως είπαμε και στην ακρόαση να αποτιμήσω το ζήτημα και θα ήθελα επομένω στην προσέγγιση σας στο πρόγραμμά σας να λάβετε υπόψη κάποια εγκάρσια πολιτική ε, να μην ε, ε, ασχοληθείτε μόνο με τον υποσυντισμό αλλά και με την διατροφική αυτάρκεια. Και ακριβώς το θέμα είναι τι γίνεται με τη γη στην Αφρική γιατί τελικά ε, ε, κάποιοι ιδιοποιούνται τη γη και ε, ιδίως στην Αφρική αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίση πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους τεχνολογική μεταφορά προς τα εκεί ούτως ώστε να υπάρχει ε, περισσότερη αποτελεσματικότητα στην ε, παραγωγή. Είναι σκανδαλώδες επίσης να έχουμε κερδοσκοπία όσον αφορά την διατροφή και για τις γυναίκες ε, συμφωνώ μια που γνωρίζω στην Αφρική και πόσο σημαντική είναι η γυναίκα για το οικονομικό γίγνεσθε έχετε την εμπιστοσύνη μας και περιμένουμε να μας παρουσιάσετε ένα σφαιρικό ευρύ σχέδιο που να τα καλύπτει όλα αυτά τα στοιχεία του προβλήματος. Η κυρία Σέρα Ροντρίγκες για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πείνα σκοτώνει παιδιά, στο Νότο αλλά και στη Νότια Ευρώπη τα παιδιά υποφέρουν από ε, υποσυτισμό. στη χώρα, στην περιοχή μου, στην Γαλλικία, ε, πολλά παιδιά υποφέρουν λόγω του υποσυτισμού. Στην Ισπανία, 60% των ανθρώπων, 60, ε, των ανθρώπων έχουν, ε, διατρέχουν τον κίνδυνο υποσυτισμού και φτώχες από ε, σε σχέση με, το, με πέρυσι. Ο κόσμος δεν μπορεί να καλλιεργήσει τη γη του. Επιβάλλονται καταστροφικές συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ε, που καταστρέφουν τους λαούς. Αν δεν αμφισβητηθούν αυτές οι πολιτικές, δεν θα λυθούν τα προβλήματα υποσυτισμού του Νότου. Αν εξακολουθηθεί η πολιτική της Τρόικα, θα εξακολουθήσει και η πείνα και ο υποσυτισμός και θα επεκταθεί και στον Βορρά. Κύριε Επίτροπε, σκοπεύετε να συνεχίσετε τις ε, πολιτικές αυτές ή θα θέσετε τέλος στις πολιτικές ε, ε, εκμετάλλευση των πολιεθνικών. Θα θέσετε τέλο στι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Θα ενημερώσετε, τις, θα αλλάξετε τις γεωργικές πολιτικές, θα τις ε, μεταβάλλετε τις, ε, έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια τροφίμων. Εάν δεν προχωρήσετε σε τέτοια μέτρα θα μείνετε στα κενά λόγια και του χρόνου θα συνεχίσουμε να μετράμε το νούμερο των, ανθρώπων που είναι υποσυτισμένοι και των ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Χόιμπουχ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίζουμε μια σημαντική έκθεση γιατί είναι ντροπή να υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που πεινάνε και πεθαίνουν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και εδώ πέρα ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μακάβαν για το ότι δεν μιλάμε μόνο για υποσυτισμό αλλά και για ελλειπή σύτηση για το ότι δεν λαμβάνουν αρκετές θερμίδες τα παιδιά για μια υγιή ανάπτυξη Χρειάζεται μια ισορροπημένη διατροφή με βιταμίνες, συχνοστοιχεία και άλλα. Όμως αυτό δεν θα το καταφέρουμε εάν συνεχίσουμε να προωθούμε τις γνωστές μονοκαλλιέργειες. Χρειάζονται συστήματα με διαφορετικά είδη ε, δημητριακών που θα περιέχουν όλες τις θρεπτικές ουσίες. Εδώ πέρα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει τις συστάσεις του ειδικού απεσταλμένου για την διατροφή που ακριβώς περιγράφει ως λύση για αυτές τις χώρες μια διαφοροποιημένη γεωργία. Η σημασία της ε, γεωργίας επίσης είναι μεγάλη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να ενισχυθούν οι μικροί αγρότες γιατί αυτοί έχουν την δυνατότητα να διαδώσουν αυτά τα συστήματα πολλαπλών καλλιεργειών που θα ανταποκρίνονται και στις τοπικές διατροφικές συνήθειες επίσης ε, και θα αναπτύξουν και την τοπική ε, οικονομία. Μετά έρχεται και η επεξεργασία των τροφίμων, η μεταφορά Όλα αυτά ακολουθούν και οι θέσεις εργασίας και το πρώτο βήμα για να φύγουν από τη φτώχεια. Χωρίς γη όμως δεν μπορούν να καλλιεργηθούν τρόφιμα. Γι' αυτό σημαίνει πως πρέπει να προστατευτούν τα παραδοσιακά δικαιώματα στη γη, η πρόσβαση στη γη για τους τοπικούς πληθυσμούς και ειδικά για τις γυναίκες. Και εδώ πέρα ο νικητής δεν μπορεί να είναι αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά πρέπει οι ντόπιοι να, είναι, ε, να κρατήσουν την γη τους και να σταματήσει η αρπαγή γης. Και αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για να καταπολεμηθεί η πείνα και η φτώχεια στις χώρες αυτές, αλλά βεβαίως δεν βοηθάνε όλες οι επενδύσεις όταν οι ιδιωτικοί επενδυτές κατ' ουσίαν διώχνουν τον κόσμο από τη γη τους για να αποκτήσουν αυτή μεγάλο περιθώριο κέρδους και παράγουν για τη διεθνή αγορά δεν χορταίνει έτσι κανένα παιδί. Πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη οι εμπορικές συμφωνίες. Και οι χώρες αυτές σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών και τις διακυμάνσεις τους και από την κερδοσκοπία των χρηματιστηρίων στα τρόφιμα τα οποία τελικά αποφασίζουν εάν ένα παιδί θα πάει για ύπνο χορτάτο ή πεινασμένο. Αυτό είναι ανήθικο και πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Η φτώχεια και η πείνα θα καταπολεμηθούν με την στήριξη των ντόπιων αγροτών για να έχουν αυτές οι χώρες μια διατροφική κυριαρχία. Χρειάζεται επίσης μια οικολογικοποίηση των συστημάτων γεωργίας να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή γιατί αυτές οι χώρες πλήττονται πρώτες. Και αυτά είναι βασικά στοιχεία στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και άμεση δημοκρατία ο κύριος Μπασίρ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε, θυμάμαι πριν από 30 χρόνια, το 1985, ο Μπομπ Γελντορφ ε, οργάνωσε εκείνο το Live Aid για να μπορέσει να βρει χρήματα, ώστε να ανακουφίσει την Αιθιοπία ε, καλείστε να εγερθείτε, να σηκωθείτε όρθιος και να απευθυνθείτε. Να ξαναρχίσω από την αρχή. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, αγαπητοί επίτροπε, θυμάμαι πριν από 30 χρόνια, το 1985, ο Μπομπ Γκέλτοφ και άλλοι οργάνωσαν το Live Aid, ούτως ώστε να βρουν χρήματα σε σχέση με τον λοιμό στην Αιθιοπία. Τώρα στην Αιθιοπία υπάρχει κίνδυνος νέου λοιμού και αυτό ε, λόγω του ελέγχου και του περιορισμού του ύδατος του Νείλου στην Αιθιοπία Κροματία. Όμως ε, οι στρατιωτικοί στην Αίγυπτο δημιουργούν προβλήματα διότι θέλουν να επιβάλλουν απικιακά δικαιώματα επί του ποταμού Νείλου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί η Αιθιοπία ε, θα έπρεπε επειδή αντιστοιχούν το 80% των υδάτων θα έπρεπε να έχει ε, αυτό το είδο του Νείλου και για τον ηλεκτρισμό αλλά και για τη γεωργία ούτως ώστε να μπορεί να δώσει ε, τρόφιμα και φαγητό στους κατοίκους της αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί να εξασφαλιστούν όλες οι χώρες της περιοχής. ένα λεπτό κύριος Μάγερ, εγγεγραμμένος βουλευτής. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παραλά εκατομμύρια παιδιά έχουν υποστηρισμό. 2,6 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο <laughs> πεθαίνουν από πείνα. Είναι τραγικό και πραγματικά μας δροπιάζει. Και βεβαίως όλα αυτά μετά οδηγούν σε πολέμους, ε, φτώχεια και τα άλλα που φαντάζεστε. Όταν τέθηκαν οι στόχοι της χιλιετίας, ε, ο υποστησμός έφτανε το 18%, τώρα έχει πέσει το 2%, ε, αλλά εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο αυτό. Βεβαίως, ε, μεγάλη σημασία εδώ πέρα οι ειδικοί αποδίδουν στην εκπαίδευση των γυναικών για να καταπολεμηθεί η παιδική θνησιμότητα. Καταπολέμηση της στόχιας επίσης σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη αναπτυξιακή συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ήβο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Παρά αυτούς τους στόχους της χιλιετίας έχουμε ένα δισεκατομμύριο συνανθρωποί οι οποίοι πάσχουν ε, και πλήσονται από αυτήν την ε, ε, άρρωσια του υποσυτισμού και βεβαίως ε, τους δίνουμε κάποια τρόφιμα αλλά δεν αλλάζει αυτό πρόκειται όπως είπε ο Πάπας Φραγκίσκος για ένα σκάνδαλο και ελπίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε το μήνυμα του Πάπα δεν μας μπήκε από να αυτή να μας βγει από το άλλο θα πρέπει να βρεθούν τρόφιμα για όλους αλλά και δικαιοσύνη για όλους και ε, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρώπη και η διεθνή κοινότητα να ε, αντιμετωπίσει τις αιτίε της φτώχειας και του λοιμού. Η συνάδελφος Μακάβαν στη κείμενό ε, αναφέρει κάποιες από αυτές τις αιτίε, αλλά δεν τις αναφέρει όλες. Θα πρέπει επομένως να ακούσουμε αυτό που είπε ο Πάπας. Πρόκειται για τον εγωισμό του ανθρώπου αυτή ότι ο κόσμος ασχολείται μόνο με το χρήμα. Κίνητρο είναι μόνο η οικονομία για κάθε ενέργεια. Όμως ο υποσυντισμός των ανηλίκων μας δείχνει το ότι θα πρέπει να τους δώσουμε κάποια αξιοπρέπεια. Ε, ακριβώς όπως γεννιέται ο άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Και θα πρέπει να δώσουμε κάποιες εγγυήσεις, να μπορεί κάποιος να αναπτυχθεί και να έχει ε, τη σωστή διατροφή α, τις πρώτες μέρες της ζωής του, αλλά και κατά την κοίηση αυτά που κάνουμε δεν αρκούν, χρειαζόμαστε μια αρκετή, μια, μια, μια επαρκή ε, αναπτυσιακή πολιτική και να υπάρχει πρόσβαση και στην παιδεία και όπου χρειάζεται. Άρα θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας. Και δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά τα 3,1 εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι αποτελεσματικό αυτό το πρόγραμμα και ότι θα εκριζώσει την πείνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε αυτήν εδώ την αίθουσα όπως θύμισαν οι συνάδελφοι, ο Πάπας Φραγκίσκος μας θύμισε ότι η Ευρώπη φέρει ιδιαίτερη ευθύνη στην καταπολέμηση της στόχης και της πείνας στον κόσμο. Το δικαίωμα στην ε, τροφή θα είναι εγγυημένο μόνο αν ασχοληθούμε με το πραγματικό του υποκείμενο, τον άνθρωπο δηλαδή που υποφέρει από τι συνέπειε τη πείνα και του υποσυτισμού. Και αυτό σημαίνει σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο να εγγυηθούμε την συνοχή ανάμεσα στι εξωτερικέ και τι εξωτερικέ πολιτικέ τη Ένωση. μείωση τη στόχη και υλοποίηση ευρωπαϊκών επιλογών σε πολιτική όπω όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η αλληλεία και η ενέργεια. Κύριε Επίτροπε, και με αυτή τη γενική προσέγγιση που θα, ε, θα μπορέσει η Ευρώπη να σηματοδοτήσει μια στροφή στι πολιτικές καταπολέμησης της στόχια, του υποστισμού των παιδιών. Και αυτές οι επιλογές θα επαναλάβουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πια να ανεχθεί σε ορισμένες φτωχέ χώρε Με τη δική μας συνενοχή υπάρχουν ε, ε, ε, γεμάτα δοχεία ενώ υπάρχουν άδειε κοιλιέ. Και αυτό επειδή οφείλεται στην εκμετάλλευση των γεών των εδαφών. λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο υποσυτισμό των παιδιών είναι μια πληγή που σκοτώνει και προκαλεί προκαλεί σοβαρές ζημιές στην ανάπτυξη των παιδιών. Θα πρέπει αυτό μακροπρόθεσμα να το αντιμετωπίσουμε. Μια καλή αναπτυξιακή πολιτική. Όλοι μίλησαν για το θέμα του νερού, των σχολείων, τη γεωργία, τη ε, τροφική ανεπάρκεια, Όλα αυτά είναι προφανή. Αλλά αν θέλουμε άμεσα αποτελέσματα, αν θέλουμε να σώσουμε παιδιά σήμερα, τότε πρέπει να αλλάξουμε πορεία και να επιτρέψουμε στην πολιτική, την αναπτυξιακή, να ιδιοποιηθεί τα αποτελέσματα τη ανθρωπιστική βοήθεια. Ξέρουμε πώ μπορούμε να μειώσουμε την παιδική θνησιμότητα. Έχει αυτό γίνει στο Σαχέλ στο πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης, χάρη στην υποστήριξη του ΕΚΟ της ΕΚΟ. Ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν σωθεί από το 2006. Με 50 δολάρια το χρόνο δίνουμε θεραπευτικά τρόφιμα έτοιμα για χρήση υπό τη μορφή φακέλου και σώνονται τα παιδιά και η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΙΕ έχουν επικυρώσει αυτή την προσέγγιση. Σας καλώ λοιπόν όλοι να σκεφτούμε ώστε η 11η ΦΕΔ να ε, λάβει υπόψη αυτή την πρακτική, να οργανώσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα ώστε τα παιδιά υποφέρουν σήμερα από υποσυτισμό αύριο να σωθούν. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Χάσεκα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε όλο τον κόσμο παράγονται τρόφιμα για να ταΐσουμε όλο τον πληθυσμό. Και όμως, απόψε ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πάνε για ύπνο πεινασμένοι. Μεταξύ των οποίων 225 εκατομμύρια παιδιά. Το κόμμα για τα ζώα το βρίσκει αυτό απαράδεκτο. Οι αιτίε όμως δεν είναι αυτές που νομίζετε. Οι αιτίε είναι η δική μας γεωργία και τα μοτίβα κατανάλωσης. Με 10 στρέμματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αρκεί όμως να μην ε, στέλνουμε τα περισσότερα φαγητά για ζωοτροφές και βιολογικά καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική, να σταματήσουν αυτά τα 330 δισεκατομμύρια γεωργικές επιδοτήσεις κάθε χρόνο, οι οποίες καταστρέφουν τη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε επίση να τρώμε τόσο κρέας. Κάθε 5 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί από πείνα. Όσο μιλούσα, δηλαδή, πέθαναν 18 παιδιά. Είναι απαράδεκτο αυτό και πρέπει να το σταματήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και Ε, συμφωνούμε και με την εισηγήτρα αλλά και με το ότι πρέπει να σταματήσουν οι γεωρικές επιδοτήσεις. Το λόγο, το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά η κυρία Χάουταλα. Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että komissio... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο υποσχετισμός ε, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι το πρόβλημα και η έλλειψη βασικών στοιχείων ε, μικροστοιχείων που περιέχουν τα τρόφιμα και που μπορεί να βλάψουν την περαιτέρω πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η Κομισιόν λαμβάνει το θέμα πολύ σοβαρά υπόψη και όπως είπε και μόλις ο, υπο, Επίτροπος μπορεί να δράσει μέσω των οργανώσεων του ΟΗΕ. Πρόκειται για ένα θέμα όπου ε, για το πρόβλημα των μονοκαλλιεργιών έχουμε εμείς οι πράσινοι υποβάλει ε, τροπολογίες πολλές ε, υπέρ μιας αγρο σε προσέγγισης γι' αυτό έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν οι καλλιέργειες και έτσι οι γυναίκες, οι μητέρες που συχνά στην Αφρική είναι στους ε, κάμπους να δώσουν πιο διαφοροποιημένη τροφή στα παιδιά τους που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτών. Θα ήθελα πρόεδρε να πιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ε, που, για το οποίο μίλησε ο Λουί Μισελ. τα ε, εδάφη ε, καταπατώνται και χρησιμοποιώνται. Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εμπορικές συμφωνίες έτσι ώστε να βεβαιωθεί το αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή οι πολυεθνικές ε, πηγαίνουν και παίρνουν, εκμεταλλεύονται μεγάλες ε, εκτάσεις τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και θα ήθελα κάτι να γίνει γι' αυτό. Μέσω της αναπτυξιακής μας πολιτικής η ΦΑΟ ανέπτυξε ε, κάποιες θελοντικές κατευθύνες γραμμές για να γίνει σχετική έρευνα και ελπίζω πως κάποια στιγμή αυτές οι κατευθύνες γραμμές θα καταστρέψουν καταστούν υποχρεωτικές ώστε να ληφθούν υπόψη καλύτερα οι ανάγκες των χωρών ε, των αναπτυσσόμενων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε η UNICEF, ο ΠΟΕ, ο ΙΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν πρόσφατα δείξει ότι η παιδική θνησιμότητα ανάμεσα στα 0 και 5 έτη έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό την τελευταία δεκαετία. Εκατομμύρια παιδιά έχουν σωθεί. Το 2013 πέθαναν ωστόσο 6,3 εκατομμύρια παιδιά. Ο υποσυτισμός είναι η πρώτη ασθένεια στον κόσμο και το 80% των παιδιών που υποφέρουν από υποσυντισμό ζουν στην ε, Νότια Ασία ή στην, Νότια, ή στην υποσαχάρια Αφρική. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρουμε καλύτερα και να στοχεύσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Και καλό τους συναδέλφους σε αυτό το κοινοβούλιο να δεχτούν την τροπολογία μας προβλέπει εξασφάλιση ε, του νερού και της ενέργειας ως ε, ε, προϋπόθεση εκ των να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να ζήσουν αυτόνομα. 17.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα, κάθε κάθε στιγμή που περνά πεθαίνουν ακόμα 12 παιδιά. Πρέπει γρήγορα να δράσουμε. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η διατροφική κατάσταση των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών είναι ένας από τους δείκτες της οικογενειακής ευημερίας και ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της επιβίωσης των παιδιών. Ο υποσυτισμός των παιδιών είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της βρεφική και παιδική θνησιμότητας μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού και κατά συνέπεια την υγεία και την παραγωγικότητα στη μετέπειτα ζωή του. είναι επίσης ένα από τα κριτήρια που ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας συνιστά για την αξιολόγηση της ισότητας στην υγεία δυστυχώ για την ευρώπη θα πρέπει να εντάξει και νέε περιοχέ υποσυτισμού που υφίστανται τα αποτελέσματα των πολιτικών λιτότητα για την αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση. αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελλάδα παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία την ώρα του μαθήματο λόγω υποσυτισμού. χιλιάδε ελληνικέ οικογένειε με μηδενικό εισόδημα λόγω ανεργία δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά του τα απαραίτητα τα παιδιά πηγαίνουν νηστικά στα σχολεία οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από το πενιχρό μισθό τους λόγω μνημονιακών περικοπών δίνουν χρήματα στα κηλικεία για να προσφέρουν διακριτικά κολατσό σε παιδιά που γνωρίζουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν. αυτά όμως από υπερηφάνεια ή και από ντροπή αρνούνται να το δεχτούν. αντί να δώσουμε την ποιότητα ζωής που αξίζει στα παιδιά μας με λάθος πολιτικές και λάθος οικονομικά μέτρα φέρνουμε χώρε τη Ευρώπη στις συνθήκες της ζωής της υποσαχάριας αφρικής. ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βέντα για δύο λεπτά. Αγαπητοί, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, είναι πρόβλημα όλοι μα στον κόσμο και αυτού πλήσει ιδιαίτερα του ανηλίκου. Πάντω, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά ε, τους στόχους του, της χιλιετίας αλλά οι υποσυντιζόμενες αντισόμενες χώρες μειώθηκαν κατά το ίμιση αλλά το πρόβλημα ακόμα υπάρχει και είναι περίπλοκο οπότε και γι' αυτό και είμαι υπέρ αυτού του κειμένου και η βασική αιτία του υποσυντισμού των ανηλίκων είναι η φτώχεια και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ασία αλλά και την υποσαχάρια Αφρική. Κατά τη UNICEF ο υποσυντισμός πλήσει 100 εκατομμύρια ανηλίκους σε όλο τον κόσμο και, έχουμε επίσης 160 εκατομμύρια τα οποία δεν αναπτύσσονται όπως θα πρέπει γιατί σταματά η σωματική ανάπτυξη σταματά η ανάπτυξη και το μυαλό από τον υποσυντισμό. δεν μπορεί να συγκεντρωθεί κάποιος δεν μπορεί να μάθει ε, Επομένω, ε, τα παιδιά αυτά έχουν καταδικαστεί να αποτύχουν στο μέλλον και δεν μπορούν να ξεφύγουν μεγαλώνοντας από αυτόν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε ε, το πώς θα γίνει αυτή η έκθεση που χτες ψήφισαμε με τόσο πλειοψηφία για το τι θα γίνει μετά το 2015 ε, και είπαμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη φτώχεια και τον υποσυντισμό. Εγώ εργάζομαι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξη και σας τονίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αμπισόμενες χώρες και να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και έτσι στο μέλλον να έχουν την αυτάρκεια. Δεν πρέπει να λέμε όχι ε, όταν μας ζητούν βοήθεια γιατί έχουμε τόσους και τόσες οικογένειες που χρειάζονται ε, βοήθεια γιατί ο υποσυντισμός είναι κάτι το πάρα πολύ και για τις έγκες μπορεί να ε, καταστρέψει, μπορεί να σταματήσει την ανάλυση του εμβρίου και επομένω θα πρέπει να δούμε πώς οι μέλους της θα μπορούν να μάθουν, θα μπορούν να έχουν καλύτερη ζωή αλλά πάντως κάθε πέντε δευτερόλεπτα από ό,τι μάθαμε πεθαίνει ένα παιδί. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Το λόγο έχει η κυρία Μίτση για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ακούσατε τι είπε ο Πάπας. Είναι απαράδεκτο τα εκατομμύρια αυτά να πεθαίνουν από πίνανο στα τραπέζια μας έχουμε τόσο φαγητό το οποίο το πετάμε. Να δούμε τι θα κάνουμε για να σταματήσει αυτή η μάστιγα. Έχουμε αυτά τα εκατομμύρια των παιδιών, αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία ε, πεινάνε. Επομένως θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σε παγκόσμια κλίμακα και τα παιδιά να έχουν αρκετό φαγητό, να έχουν ισορροπημένη δίαιτα, αλλά και οι έγκυες ε, πλήσονται από πείνα και αυτό έχει τρομερές συνέπειες για το έμβριο. Και επίσης ε, τις ε, πρώτες μέρες ε, στη ζωή κάποιου είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή διατροφή για την ανάπτυξη και επομένω θα πρέπει να βρούμε τον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη, να βελτιωθεί έτσι η κατάσταση. Θα πρέπει επίσης στα πλαίσια της παιδείας να υπάρχει διδασκαλία για το ποια είναι η σωστή ισορροπημένη διατροφή. Έτσι θα μπορεί ο κόσμος να ζει με αξιοπρέπεια. Πρόκειται για επένδυση στο μέλλον μας. Ε, να βοηθήσουμε και τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ε, προγραμματίζει, τι θα κάνει. Πώς θα σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος της φτώχειας και της πείνας. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μπεσέρα Βαστερετσέα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μάκαβον για την εξαιρετική σας έκθεση. Ε, μιλούμε ε, για το τι γίνεται για, για, για τους ανηλίκους μας όσον αφορά την ε, φτώχεια σε μεγάλες χώρες αλλά σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα όταν λέμε για αυτά τα τρία εκατομμύρια των παιδιών που κάθε μέρα δεν έχουν αρκετό φαγητό το επονίδιστο και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τους δώσουμε τα, τα, προσόντα, και τα, το, τα τρόφιμα για να γίνουν πολίτες σαν όλους αυτά τα παιδιά. Να βάλουμε ένα τέρμα στην πείνα στις αντισόμενες χώρες. Και επίσης να η πείνα στους φτωχούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βοηθήσουμε και στο επίπεδο της Γεωργίας στις αντισόμενες χώρες. Έτσι θα υπάρχει αξιοπρέπεια, θα υπάρχει ε, ασφάλεια διατροφική και η κοινωνία θα πρέπει να σκεφτεί το μέλλον των ανηλίκων. Είναι υποχρεωσή μας να αναλάβουμε δράση τώρα και επομένως θα πρέπει να, δούμε, να βοηθήσουμε και τους ανήλικους αλλά και τους ενήλικους. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε αυτό το που θέλουμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην διατροφή. Αυτό είναι ηθική υποχρέωση και έχουμε όλους αυτούς τους ανηλίκους κάτω από πέντε ετών που πλήσονται και έχουμε ε, αυτούς που έχουν αυτή την καχεξία και οπότε θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι πρόκειται για κάποια αναγκαιότητα, κάτι το οποίο πιέζει. Θα πρέπει μένως ταχαίως να λάβουμε μια πρωτοβολία αυτή που συζητούμε σήμερα. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ε, την Τρίτη ψηφίσαμε ε, μεγάλη πλειοψηφία είπαμε να γίνει ένα ψήφισμα όσον αφορά το πρόβλημα αυτό και να γίνει αυτό το 2015. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να γίνει και θεωρούμε ότι η διατροφή είναι βασικό δικαίωμα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μηδενική πίνα στόχος αυτός έχει τεθεί με το 2025 να εκριζώσουμε και την πείνα και τον υποσυντισμό και να, έχουμε, να μην έχουμε πια και αυτή την κρυφή πείνα που πλήσει τους ανηλίκους και τις γυναίκες όταν θυλάζουν οπότε θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε και με τις, ε, ε, και στο πλαίσιο του ΟΗΕ να καταπολεμήσουμε τον υποσυντισμό. Έχουμε εδώ πέρα το πρόγραμμα για το 2030 και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα εκριζώσουμε αυτήν την, ε, την πείνα που πλήσει τους ανηλίκους και άρα θα πρέπει να υπάρχει σαν τις χώρε χώρες νερό, θα πρέπει να υπάρχει βιώσιμη γεωργία, ε, να έχουμε ένα υγιεινό περιβάλλον, να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες επίσης και όλη την οικογένεια εκεί που πλήσετε και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια καλύτερη διαχείριση της γης της χώρας αυτής. Ο κύριος Ταραμπέλα για 1,5 λεπτό. Monsieur monsieur... le Président, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως μέλος ε, της Επιτροπής των Γυναικών και των Δικαιωμάτων των Γυναικών θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μέσα στην αδικία που πλήττει τα παιδιά που πάσουν από υποσυτισμό έχουμε τα, τα κορίτσια τα οποία ε, ε τρεις περισσότερες φορές ε, διατρέχουν τον κίνδυνο να υποφέρουν από σοβαρό υποσυτισμό. Είναι ακόμα πιο ευάλωτα απέναντι στα, στα, προβλήματα της ανάπτυξης και συχνά πεθαίνουν πολύ μικρά ε, πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πολιτιστικά και θρησκευτικά εμπόδια σε αυτές τις ε, συμπεριφορές που, που, επιβαρύνουν τα κορίτσια και να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Επιπλέον στις συστάσεις ε, του ΟΗΕ βλέπουμε ότι αν οι γυναίκες γεωργοί είχαν τα ίδια μέσα πρόσβαση στα ίδια μέσα όπως οι άνδρες γεωργοί θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά τρεις φορές τη γεωργική παραγωγή. Δηλαδή 100 με 150 εκατομμύρια κόσμος θα γλίτωνε από την πείνα. Οι ανισότητες στη στα κορίτσια και στα χώρια από την πολύ μικρή ηλικία θα βελτίωνε τις προπτικές των γυναικών γεωργών καθώς και την, θα βοηθούσε στην καταπολέμηση της, του υποσυτισμού στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες και νομίζω είναι προτεραιότητα. Ε, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από πείνα. 2,6 εκατομμύρια παιδιά στι αναψώμενε χώρε πεθαίνουν κάθε χρόνο από υποσυτισμό. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2014 500.000 άνθρωποι θα έχουν υποσυτισμό και οι λόγοι διαφέρουν. Πολλοί από αυτούς είναι ανθρωπογενείς, άρα μπορούν να αποφευθούν. Συχνά μιλάμε για συγκρούσεις, ε, πολιτική αστάθεια, όλα αυτά προκαλούν ε, την, ε, τον υποστηρισμό των παιδιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα στατιστικά δεδομένα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα αποτελέσματα των πολέμων σε παιδιά. Οι λοιπόν πρέπει να φροντίσουν περισσότερο για τον επισητισμό των παιδιών τους και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινητοποιήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα αυτών και να συνεργαστούν με τρόπο αποτελεσματικό με τους διεθνείς φορείς. Οι πόροι, οι οικονομικοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, όμως σε πολλές περιπτώσεις όπως το Μαλί ας πούμε ή τη Συρία ε, το καλύτερο μπορεί να γίνει να σταματήσει ο πόλεμος και να δημιουργηθεί ένα πολιτικά σταθερό περιβάλλον χάρη σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Ε, κάτι τέτοιο είναι εξίσου σημαντικό. Ευχαριστώ. Κύριος Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο υποσυντισμό των παιδιών και η πείνα στον κόσμο θα πρέπει να είναι πραγματική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν οφείλει να εκπονήσει σοβαρέ πολιτικέ κατά των, ε, ε, της πατάλης των τροφίμων. 225 εκατομμύρια είναι τα παιδιά που υποφέρουν από τον υποσυτισμό και από καθυστέρηση της ανάπτυξής τους. 26 εκατομμύρια παιδιά δεν πεθαίνουν κάθε χρόνο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καλείται να επιτείνει τις προσπάθειές της για αυτό το θέμα. Η περιπλοκότητα της προσέγγισης θα έπρεπε ε, να οδηγεί σε δημιουργία ενός στρατηγίου που να μπορεί να κατευθύνει διάφορες δράσεις ολοκληρωμένες ώστε να καταπολεμηθεί και να εκριζωθεί αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καλείται και θα πρέπει να σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, τον G8 τις, τις χώρες να μπορέσουν λιγότερο εγωιστικά, να μπορέσουν να βάλουν ε, τις εταιρείες ε, ε, τις βιομηχανίες μάλλον του γεωργικού τομέα να αναπτύξουν επαρκή τρόφιμα και διατροφή για όλο αυτό το κόσμο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πριν από 70 χρόνια μία χιλιανή είπε ότι είμαστε ένοχοι, έχουμε κάνει πολλά λάθη, αλλά το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά στην απαρχή της ζωής τους. Και πολλά θα πρέπει να γίνουν, πολλά μπορούν να περιμένουν, αλλά όχι οι ανάγκες των παιδιών δεν περιμένουν, γιατί θα πρέπει να μπορούν να αναπτυχθούν ε, όταν γεννώνται πρέπει να αναπτυχθούν γιατί τα κόκαλα, η ιστή, όλα ε, αυτό πρέπει να γίνει σήμερα τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει όλοι είμαστε υπεύθυνοι η Ευρώπη είναι ένοχη κύριε Στυλιανίτη σας ευχαριστούμε για τα όσα είπατε και νομίζω ότι έχετε δεσμευτεί ότι σας ενδιαφέρει το θέμα και θα προχωρήσετε σε μια προσπάθεια συντονισμού και ότι θα πρέπει να γίνει συντονισμό τη ε, εσωτερική και τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο να ενεργήσουμε με τρόπο ισορροπημένο. Επίσης μου φαίνεται πάρα πολύ σωστή αυτή η αξιολόγηση των επιπτώσεων που είπατε ότι θα γίνει και θα την κάνετε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Κυρία Μακάμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κείμενό σας, είναι σημαντικό το θέμα, οπότε ε, είδαμε ότι την Τρίτη ε, ε, εγκρίναμε την προσπάθεια αυτή που θα γίνει για το 2015 και μετά για αυτό το, το, το πλαίσιο πολιτικής που θα υπάρχει, το, πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο και Ελπίζουμε ότι κάτι θα πετύχουμε γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και αυτά τα οποία είπε ο Πάπας κατά την επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο. Τι είπε. Είπε ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη ούτε στην Ευρώπη ούτε πουθενά όταν έχουμε την σπατάλη τέτοιων και τόσο μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων. Μην το ξεχνούμε αυτό το οποίο είπε. Είπαμε ότι εν μέρει πετύχαμε και από τους στόχους του, της χιλιετίας, αλλά ακόμα μένουν πολλά να κάνουμε, όχι άλλα λόγια, αλλά δράση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα θέλω να αρχίσω με το να αναγνωρίσουμε το ότι έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βοηθήσει για τους ανηλίκους. Βέβαια, ε, είδαμε ότι όλο ένα και μεγαλώνει το πρόβλημα αυτό το οποίο έχουμε ε, και αυτό εμποδίζει την ανάπτυξη. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δώσει όλα αυτά τα χρήματα, αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειε. και επομένω θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει όλα αυτά να τα εντάξουμε σε κάποιο πλαίσιο για να μπορέσουμε να καλύψουμε ε, τους ε, στόχους μας, αυτά τα οποία έχει θέσει ο στόχο και η UNICEF. Και επομένω θα πρέπει να δούμε τρει βασικού στόχου, στόχους. Πρώτα-πρώτα τι θα γίνει για το παιδί τι πρώτες χίλιε μέρες της ζωής. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αυτό και σημαντικό για την ανάπτυξη. Πώς θα βοηθήσουμε τους μικροκαλλιεργητές και επίσης που είναι σημαντικό να βοηθήσουμε στην συμμετοχή των ε, γυναικών. Ε, όπως ξέρουμε, ε, κάνει πολλά στην οικογένεια η γυναίκα, οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε να, συμμετέχει στη διαχείριση των υγειών και η γυναίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 3,1 ε, είπαμε ότι είναι αυτά τα εκατομμύρια για τις παρεμβάσεις αλλά επίσης είπαμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη θνησιμότητα των παιδιών κάτω από 5 λόγω του υποσυτισμού. Από αυτό είναι επομένως ένας βασικός στόχος της χιλιετίας. Και όταν λέμε για υποσυντισμό, αυτό πάντοτε έχει να κάνει και με την διατροφική ασφάλεια και με την φτώχεια. Αλλά ε, το θα πρέπει να δούμε για το πώς θα υπάρχει περισσότερη υγιεινή στο, στην οικογένεια, στο νοικοκυριό και αν υπάρχει καλύτερη ε, προσβασιμότητα τη υπηρεσία υγεία 250 εκατομμύρια. Τώρα δεν έχουν όμω υγιεινέ συνεχεί διατροφέ και κυρίω αυτό γίνεται στην Αφρική, στην Ασία και στην υπόσαχαρη Αφρική. Ένα στου ε, νέα ανθρώπου στον κόσμο βρίσκεται τέτοια κατάσταση. Επίση έχουμε 66 εκατομμύρια ε, ανηλίκου ε, οι οποίοι πάνε σχολείο και πεινάνε. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικέ οι πρώτε χίλιε μέρε τη ζωή για να αναπτυχθεί καλά ένα ανήλικο ε, και, να μεγαλώσει το πάντων με αξιοπρέπεια. Επομένω τα πράγματα είναι σε κρίσιμο σημείο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τον υποσυντισμό. Επίση, είναι αλήθεια ότι κατέβαλε προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να καινοτομήσουμε, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μακρόπνο, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν δεν υπάρχουν ε, τα τρόφιμα, θα πρέπει να υπάρχει όμως και όταν υπάρχουν, και όταν υπάρχουν τρόφιμα να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, να κάνουμε περισσότερα για υγεία, για παιδεία και για την ισότητα των ευκαιριών. Οι γυναίκε που ασχολούνται με τη γεωργία, εάν είχαν τα ίδια δικαιώματα, εάν είχαν τι ίδιε ευκαιρίε, εάν είχαν την ίδια προσβασιμότητα στι σχετικέ υπηρεσίε με του άντρε, ε, αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Δεν θα πίναγαν ούτε οι γυναίκε αυτέ, ούτε τα παιδιά. Άρα θα πρέπει ε, να εξωθήσουμε την Επιτροπή και, και τους Επιτρόπους να κάνουν περισσότερα, να επενδύσουμε σε προσπάθειες σε αυτό τον τομέα. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα παρά να μιλήσω για τον υποσυτισμό, να μιλήσω για την πείνα στις αναπτυσσόμενες χώρες πείνα των παιδιών όμως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στις χώρες ε, των μνημονίων όπου έχει παρεμβεί η Τρόικα. Έχει προκληθεί πείνα από την ανεργία και από την αποσία κράτους. Στη χώρα μου την Πορτογαλία τα σχολεία εξασφαλίζουν ένα ζεστό ε, φαγητό για τα παιδιά. Είναι ανοιχτά Σάββατα και Κυριακές για να εγγυηθούν ότι τα παιδιά δεν θα μείνουν ε, νηστικά. Και ξέρετε γιατί. Γιατί σε μια χώρα ανεργίας και αναγκαστικής μετανάστευσης οι ε, γονεί δεν έχουν πώς να θρέψουν τα παιδιά τους. Το 2011, στο απόγειο της κρίσης, το 30% των παιδιών της Πορτογαλίας είχαν πέσει στη φτώχεια. 35.000 παιδιά υπολογίζουμε ότι πεινάνε στην ε, χώρα μου. Η πείνα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Τι θα κάνει η Κομισιόν σε σχέση με τη φτώχεια και την πείνα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χέις για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και πραγματικά καλοδεχούμενο αυτό το ψήφισμα και να συγχαρώ και την κυρία Μακάβαν για τη δουλειά που έκανε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχει σημαντική πρόοδο στον τομέα του υποσυτισμού τα τελευταία χρόνια και καθώς περνάμε στο 2015 όχι μόνο όσον αφορά τους στόχους της χιλιετίας, αλλά και στο βάρος που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς είναι Ευρωπαϊκό έτος της ανάπτυξης, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα εντός της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για να σημειωθεί πρόοδος. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κάθε μέρα που περνά 20.000 παιδιά πεθαίνουν από υποστηρισμό 90% στην Ασία και την Αφρική. Μπορούμε να προλάβουμε όλους αυτούς τους θανάτους και πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Άπαξ και διαπαντός. Πρέπει οι πανεσυνάδελφοι να στηριχθούν οι αγρότες στις χώρες αυτές, να έχουν το σωστό εξοπλισμό. Μιλήσαμε επίσης για την ανάγκη να βελτιώσουμε τη διατροφή για να υπάρχει η σωστή ε, παροχή τροφίμων και ειδικά να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις ε, κατά των γυναικών και τη θέση τους βεβαίως στη δουλειά και στο σπίτι. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τον θυλασμό για να μην υπάρχει πρόβλημα με τα μολυσμένα νερά και πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο γύρω από τις πρώτες χίλιες μέρες των παιδιών. Τα πρώτα δύο χρόνια έχουν κρίσιμη σημασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η κινητικότητα των ε, τιμών των τροφίμων είναι ένα άλλο ζήτημα και η ασφάλεια των τιμών των τροφίμων. Έχουν γίνει πολλά και μπορούν να γίνουν περισσότερα και αν αποφασίσουμε να το κάνουμε από κοινού με τους εταίρους μας παγκοσμίω, μπορούμε νομίζω να το λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δεχτεί αιτήματα από οκτώ συναδέλφους. Ε, μπορούμε να μιλήσουν όλοι, αλλά ζητώ να τηρήσουν όλοι το όριο του ενός λεπτού που προβλέπει ο κανονισμός, έτσι ώστε να μην ε, λείψει χρόνος και να μιλήσουν όλοι. Παρακαλώ τον κύριο Γλέζο για ένα λεπτό. Ο τίτλος του θέματος ο υποσιτισμός των παιδιών αποτελεί μια αποκαλυπτική ομολογία. παραδεχόμαστε δηλαδή όλοι ότι υπάρχει υποσιτισμός στα παιδιά. όσα ακούστηκαν όλες οι διαπιστώσεις είναι σωστές. όμως δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. πρέπει να φτάσουμε στην αιτία. για ποιο λόγο δημιουργείται το φαινόμενο του υποσιτισμού ιδιαίτερα στα παιδιά αιτία είναι το σύστημα που έχει θεό του το χρήμα. Ας μην εθελοτυφλούμε. Το κεφαλοκρατικό καθεστώς, το παγκόσμιο αυταρχικό καθεστώς, η G8 Παύλα 20, το καθεστώς των πολέμων εναντίον λαών εθνών πολιτών, το καθεστώς κατασκευής όπλων και του εμπορίου των όπλων και μου έκανε εντύπωση γιατί εχθές ο δεν σε μια εκστρατεία εναντίον της κατάργησης των όπλων. Ο ενεργός πληθυσμός, αναφέρουν οι επιστήμονες, εάν δεν υπήρχε το προηγούμενο καθεστώς δεν θα χρειαζόταν να δουλεύει μονάχα ένα λεπτό την ημέρα για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και να εξαλείψει τον κανονισμό, το, το καθεστώς αυτό. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, τα νούμερα τα ακούσατε, πάνω από 800, ε, πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι υποστήριζονται παγκοσμίω. Ε, εγκρίθηκε και το ψήφισμα της Ρώμης ε, για την καταπολέμηση του υποσυτισμού ως ε, συμπρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τους στόχους χιλιετίας η Ουγγαρία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη στρατηγική αυτή μέχρι το 2025 ο αριθμός ε, των παιδιών που υποσυτίζονται πρέπει να μειωθεί κατά 40% παγκοσμίω. Προκλήσεις αυτές για όλους μας. Θέλω εδώ πέρα να σας πω πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ήδη κάποιες καλές πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Ας δούμε παραδείγματος χάρη το ουγγρικό πρόγραμμα που λέγεται Υγιεινή Διατροφή για τα Παιδιά. Αν διαδοθεί αυτή η πρακτική αυτό θα μας ωφελήσει όλους εντός και εκτός της Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, σημερινή συζήτηση ακούσαμε πάρα πολλά νούμερα. Εγώ ένα νούμερο μπορώ να στηρίξω, το 0. Δεν μπορεί να λέμε 40 και 50%. Ο στόχος πρέπει να είναι 0. Αν είναι τόσο σημαντικό για όλους μας ε, οι πρώτες χίλιες ημέρες των παιδιών να είναι υγιείς τότε η Κομισιόν έχει την αποστολή να μειώσει τον αριθμό αυτών ε, στην Ευρώπη πρώτα στο μηδέν. Στην πατρίδα μου, στην Ουγγαρία, ένα στα δύο ε, νεογέννητα αντιμετωπίζει την προοπτική της πείνας. Δεν είναι δυνατόν μόνο να κάνουμε τον έξυπνο στους άλλους, να δούμε και τα δικά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ θα ήθελα να σας πω πως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για τα παιδιά που ζουν στα στρατόπεδα προσφύγων. Ανά τον κόσμο υπάρχουν όλο και περισσότεροι πρόσφυγες και δεν λύνει εγκαίρως το πρόβλημα η διεθνής ε, κοινότητα. Το πρόβλημα αυτών των παιδιών λοιπόν επιδεινώνεται συνεχώς και υπάρχουν όλο και λιγότερα μέσα για να καταπολεμηθεί. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει μόνο να βοηθάει ε, αυτούς που έχουν ανάγκη αλλά να συνεισφέρει στον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο και πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει ακόμα χρόνος. Κύριε Πρόεδρε, ο υποσυτισμός των παιδιών εξαπλώνεται ραγδαία καθώς αυξάνεται η παγκόσμια φτώχεια. Ο υποσυτισμός λόγω της μερκελικής λιτότητας πλήττει πλέον και τα παιδιά του ευρωπαϊκού νότου. στην ελλάδα η τρόικα και τα μνημόνια έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. το 40 του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας και οι άνεργοι έχουν φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο. σύμφωνα με τη unicef πάνω από 439.000 παιδιά ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. η παιδική φτώχεια έφτασε το 2012 στο 40,5% και η κατάσταση είναι τραγική ιδιαίτερα στις πολύτεκνες οικογένειες. Τα περιστατικά με λιποθυμίες των παιδιών στα ελληνικά σχολεία λόγω πείνας είναι συχνά. Μόνη λύση κύριε Επίτροπε είναι η κατάργηση των μνημονίων και η ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω για τη ρίζα του κακού, για τις αιτίες της στόχιας στις εμπισόμενες χώρες. Κάποιες από αυτές τις αιτίες έχουν αναφερθεί σήμερα αλλά όμως βεβαίως είναι και ο πόλεμος μια είναι το έγκλημα, είναι το οργανωμένο έγκλημα γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές βέβαια και στην Ευρώπη που υποστηρίζουν τα παιδιά ας πούμε στην Ανατολική Ουκρανία εκεί τα παιδιά υποφέρουν είναι ανήκουστα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί ανήκουστα για ε, τον πολιτισμό μας βέβαια έχει κάνει ε, κάποια πράγματα η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει ειρήνη, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να κάνουμε κάτι για το πρόβλημα βεβαίω και συμφωνώ με όλα όσα είπε η συγγήτρια για όλε αυτέ τι ε, δράσει. Αυτό το οποίο χρειάζεται όμω να υπάρξει ειρήνη, να υπάρξει συνεργασία ε, παντού στον κόσμο. Οπότε το πρόβλημα αυτό θα είχε αντιμετωπιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παράδειγμα προ ε, μίμηση. Το είπε αυτό και ο Πάπα Φραγκίσκο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πείνα και ο υποσυντισμός των παιδιών έχουν διαρθρωτική ε, διάσταση και πολύ συγκεκριμένα αίτια, όπως η ευνόηση του μοντέλου του αγροβιομηχανικού με την ε, ε, αύξηση την ποσοτική του αγροτροφημικού τομέα παγκοσμίω. Έτσι όλα αυτά γίνονται εις βάρος των μικρομεσαίων γεωρικών εκμεταλλεύσεων που εξασφαλίζει το 70% όμως ε, της ε, τροφής για τις ε, φτωχές τάξεις του πλανήτη. Η εμπορευματοποίηση είχαν και έχουν ως, έχει ως αποτέλεσμα, την εγκατάλειψη της καλλιέργειας των εδαφών, την εξάρτηση των πολλών και την, από τους λίγους. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι άδικο, καταπιεστικό και γι' αυτό και ιστορικά έχει καταδικαστεί. Είναι λυπηρό, αλλά πρόκειται για ένα ηρεμιστικό, είναι, είναι, είναι πραγματικά ε, λυπηρό το ότι προσεγγίζουμε αυτό εδώ το θέμα ε, με αυτόν τον τρόπο. Ο, ε, η καταπολέμηση του υποσυτισμού των παιδιών είναι θέμα ηθικό και είναι και θέμα δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Με τη διαδικασία του Κάτσου κυρία Γιακονσάρη.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 αυτό το ψήφισμα είναι εξαιρετική σημασία και μάλιστα αποτελεί ένα βήμα μπροστά ε, στον αγώνα κατά του υποσυτισμού των παιδιών και είναι ζωτική σημασία. Θα ήθελα να θέσω την ίδια ερώτηση όπως ο συνάδελφος Κλέγκος. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο, γιατί έχουν γίνει πολλές αναλύσεις επ' αυτού, αλλά εγώ θα ήθελα να συμβάλλω επίσης. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό στην Αφρική είναι αυτό το θέμα της αρπαγής ε, της γης οι πλούσιες αραβικές χώρες και οι πολυεθνικές εταιρείες αγοράζουν τη γη για δυο ψίχουλα γιατί γνωρίζουν πως ο πλανήτης δεν μπορεί να μεγαλώσει και έτσι πιάνουν την καλλιεργήσιμη γη ε, και όταν γίνονται ιδιοκτήτες αυτής της γης μπορούν να αποφασίσουν τι θα παραχθεί και σε ποιες ποσότητες. Έτσι τα μικρά ε, οι μικρές εκμεταλλεύσεις υποφέρουν, πράγμα που οδηγεί στη διάλυση του γεωργικού τομέα στην Αφρική. Δεν είναι αυτό νεοαπικιοκρατία. Εγώ θα έλεγα πως ναι, η Κομισιόν θα πρέπει να εστιάσει πολύ περισσότερο την προσοχή όταν πρόκειται για την αρπαγή των γεών. Ευχαριστώ. Μάικρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή για τις ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούστηκαν παραδείγματος χάρη τον ρόλο των γυναικών των ε, ντόπιων αγροτών και βεβαίως το θέμα της ε, εγγύου ιδιοκτησίας Υπάρχουν ε, πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα εδώ πέρα. Νομίζω πως ε, η επιτάχυνση των ε, πρωτοβουλειών επιβεβαιώνει πως η Κομισιόν είχε δίκιο όταν έθεσε την διατροφή ως πρώτη προτεραιότητα της ανάπτυξης. Τα κράτη-μέλη έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για το σχέδιο δράσης και η Ιταλική Προεδρία προετοιμάζει συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτό θα αυξήσει βεβαίως ε, την, ε, τον συντονισμό και την δέσμευση των κρατών μελών και θα επαναβεβαιώσει τον ηγετικό ρόλο της Ένωσης την προηγούμενη εβδομάδα η διεθνής διάσκεψη έδειξε πως η πρόθεση άνω των 170 εκπροσώπων κρατών ε, για την ε, υιοθέτηση της Ρώμης ήταν ένα καλό σημάδι και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως καλωσορίζω το αίτημα για ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διατροφή και την πρωτοβουλία της κυρίας Μακάβαν, πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης. Και ελπίζω οι κοινέ μας προσπάθειες να στείλουν πια τον υποσυντισμό στα βιβλία της ιστορίας για να ανοίξει ο δρόμος της βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή τη συζήτηση, για αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Η συζήτηση για το θέμα αυτό έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση της συζήτησης. Η ψηφοφορία θα, δια... θα διεξαχθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στις συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου με διάρκεια μία ώρα κατά νότατο όριο σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού.